Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να αρχίσουμε, έχουμε ψηφοφορίες. Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε πώς πάνε οι κάρτες. Okay. Oui, pardon.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 Έτσι. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. 6 δηλαδή λέει εδώ. 6. Συμβιβαστική υπέρ. Είναι το κείμενο του κυρίου Κοράου. Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. η συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Το ΕΛΚ να ψηφίσει παρακαλώ. Δεν έχει κατάλογο ψηφοφορίας. Το κείμενο του κυρίου Κοράου. Λοιπόν, πάμε. Συμβιβαστική έξι στην έκθεση Κοράου. Υπέρ. Κατά. Abstention adoptée. Αποχές εγκρίνεται. Amendement 27. Η τροπολογία υπαριθμών 27 είναι από κάτω ακριβώς. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 36. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 9. συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε παρακαλώ. Η συμβαστική 23 άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε, παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Λοιπόν, η συμβιβαστική η τροπολογία 23 επαληθεύεται ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Bon. Amendement 45. Η τροπολογία 45. Πάμε, Είπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, νομίζω. Νόιζερ υπέρισε, μάλιστα, εγκρίνεται. 46. Είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 47. Όχι. Προχωρούμε. Καταπέπτουν, καταπέπτουν συγγνώμη. 11 συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. Καλώς. 78. αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ισοψηφία 12-12, αλλά απορρίπτεται παρόλα αυτά. Η τροπολογία συμβαστική 14. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 92 τροπολογία υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Είμαστε στην 92. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική απορρίφευση για την τροπολογία 92. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, όχι, απορρίπτεται, ισοψηφία. Όχι, 13-11 είναι. 13-11. Εγκρίνεται. 93 υπέρ πώς είπατε 93 Συγγνώμη πρόεδρε Κάποιος δεν ψηφίζει ηλεκτρονικά Άλλο λέτε, άλλο μας βγαίνει ε, στην οθόνη. Κάποιος δεν έχει την κάρτα του. Γι' αυτό σας το λέω. Α, κάποιος δεν έχει την κάρτα του. Ναι, αγαπητοί συνάδελφε. Ο συνάδελφος Βέντα έχει ξεχάσει την κάρτα του και ψηφίζει διανατάσεως της χειρός και κάθε φορά μετράμε την ψήφο του αναλόγως. Γι' αυτό βλέπετε. Να έρχεστε με κάρτα. Έτσι, έτσι. Ναι. No card, no vote. Καλά. Ευχαριστώ. Pour. Contre. Abstention. Adopté. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβιβαστική 16. Ορίστε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 93 είμαστε. Πάμε πάλι 93 και επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ο κύριος Μέντα είναι υπέρ. Είναι 12-11. Συμβαστική 16. Σας παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, παλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαρθμών 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία έτσι. Συμβαστική 17 17, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Μου λέγουν ότι εδώ οι τροπολογίες 109, 110 και 111 καλύπτονται. Υπέρ τη 18 λοιπόν συμβαστική Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ο κύριος Βέντα έκτισε κάρτα. 11, 11. Όχι, όχι, δεν είναι ισοψηφία, είναι 11-10. Έχει κάρτα κύριο Βέντα και ψηφίζει με την κάρτα. Εγκρίνεται ah, λοιπόν. 11-10. Η κυρία Χάουταλα ζητεί το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν ψηφίσαμε οι δυο μας. Μπορείτε να μας ε, διευκρινίσετε τι ψηφίζαμε τώρα. Τη συμβαστική 18 ε, τότε δύο ε, ψήφους των πρασίνων υπέρ. Εντάξει, εγκρίθηκε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ωραία. Ωραία, ευχαριστώ. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Η τροπολογία 137 ειπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 του προπολογισμού ειπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 ειπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 και 21 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι αιτιολογικές αναφορές έχουμε την τροπολογία ε, που λέγεται συμβιβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ φωνές από κάτω. Είναι η τροπολογία 8. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Le vote est clos. Pérez. Εγκρίνεται. Le vote final. Le vote final. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Και ονομαστικά επίσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν το χαμηλώσω γιατί... Τεκλού. Πέρας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ. 0 κατά και 4 αποχές. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Φροντζούλικα, από όλου τους συναδέλφους, όταν σας ζήτησα να το ελέγξετε, αλλά έχω την εντύπωση ότι το ΕΛΚ καταψήφισε, γιατί δεν βλέπω τι γίνεται από πίσω μου, και ο φίλος μου από τη Ρουμανία, κύριος Πρέντα, νομίζω ότι ζήτησε να ψηφίσουν κατά. Ζητώ συγγνώμη που σας ζήτησα επαλήθευση και τελικά ήταν ομόφωνα υπέρ το αποτέλεσμα. Η κυρία Χάουταλα. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω το εξή. Οι δυο μας εδώ ψηφίσαμε αποχή οι πράσινοι. Όχι ότι δεν ήταν καλή οι συμβιβασμοί, παρά ήταν συμβιβασμοί. Και αν διαβάσετε το κείμενο, έχουμε πολλές επαναλήψεις, σχεδόν όλες οι τροπολογίες έχουν μπει σε συμβιβαστικές. Το κείμενο δεν είναι πάρα πολύ συνεκτικό και θα ήλπιζα να, είχαν, να έχουν συζήτηση και ηγητές πριν πάει στην Ολομέλεια η έκθεση για να σβηστούν κάποιες επαναλήψεις και κάποια στοιχεία που δεν έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Δηλαδή παρά είναι συμβιβασμός. Είπαμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό, αλλά έχει γίνει σούπα τώρα εδώ πέρα. Θα συνεχίσουμε τώρα τις ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε επί προφορικής ερωτήσεως. Είστε έτοιμοι? Προφορική ερώτηση λοιπόν. Παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι συμβαίνει, λέει ο πρόεδρος, συμβαίνει κάτι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα.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 Ωραία, κάνουμε τώρα την τελική ε, ψηφοφορία, η τελευταία, η τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Πολύ ωραία, εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ. Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Αρχίζουμε λοιπόν. Προφορική τροπολογία 4. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά 57 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 58 θα το κάνουμε, το ψηφίζουμε μαζί με το, 25, μαζί με το 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές ε, επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία επαλήθευση επί της τροπολογίας 60 εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι θα κάνουμε και εδώ επαλήθευση για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64. 64 λέγω. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 75 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79. Α, 78. Ψηφίζουμε το 78. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Την 79 ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές ε, επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. 82 καταθμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 ε, υπέρ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 88 υπέρ 87 μάλλον 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση επί της τροπολογίας 90. Πολύ ωραία. Επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 95. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80-96. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 και 99 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100, 100, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 101, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 την ψηφίζουμε. Α, 108 και 114 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110 δεν ψηφίζουμε. Ε, ψηφίζουμε την 111 υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση παρακαλώ επί της τροπολογίας 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 112 καταπίπτει. Όχι, την ψηφίζουμε. Τροπολογία 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116. Όχι. Και αυτή καταπίπτει. Τροπολογία 16. Ναι, τροπολογία 16 στην αιτιολογική αναφορά A. Ναι. Αιτιολογική σκέψη, συγγνώμη. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Επί της τροπολογίας 19. 19. Επαλήθευση για την τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 21 και 22 μαζί υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 <coughs> υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται 25 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση από τις 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Όχι, τροπολογία 31. Το 30 δεν το ψηφίζουμε. Όχι, την ψηφίζουμε και την 30. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ μαζί με την 34 γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πηγαίνουμε στην τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ο προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ. Στροπολογία 43. Επαλήθευση επί της τροπολογίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται λέει ο Πρόεδρος. Διορθώνει. Τροπολογία 50 απερίφθη. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι αιτιολογικές αναφορές τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, περνάμε τώρα στον, στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, υπέρ της 6 κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε on block από την τροπολογία 8 μέχρι την 13. 8 με 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του, του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ.